Ακολουθούν τώρα οι επεξηγήσεις ψήφου. 50... Uh, επεξηγήσεις έχουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορο, θα είμαι αυστηρό, θα σας διακόπτω, θα σας παίρνω το μικρόφωνο. Συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Η έκθεση για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων Συνόδου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2012. Ο κύριος Μπάτεν για ένα λεπτό. Very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία επεξήγηση θέλω να κάνω για το χρονοδιάγραμμα του 2012. Ε, φυσικά είναι ανοησίες και τίποτε άλλο αυτά που ψηφίσαμε, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα με τα τρία κοινοβούλια, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο. Όλοι το ξεχνάνε το Λουξεμβούργο. Το συνολικό κόστος ε, είναι 250 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, αν δεν κάνω λάθος θα ήθελα να κάνω μια επικοδομητική αντιπρόταση. Αντί να συνεδριάζουμε 12 φορές ε, στο Στρασβούργο, γιατί δεν κάνουμε 12 συνόδους ε, στο Στρασβούργο μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή τρεις ε, συνεδριάσεις την ημέρα, έτσι, για αυτή τη βδομάδα για να μην περνάμε όλη την ώρα μας εδώ, να είμαστε στις Βρυξέλλες και να εξοικονομούμε χρήματα και δεν θα χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε. Ο κύριος Χάνεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, είναι φοβερό που ερχόμαστε και προσκυνάμε εδώ κάθε μήνα και αλλάζουμε έδρα. Ε, ε, εκατομμύρια χαλάμε σε αυτό και Επίσης, επειδή μεταφέρονται όλοι με φορτηγά, με αυτοκίνητα, επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εντάξει, τα ξέρω τα περί συμβολικής σημασίας, ιστορικής σημασίας του Στρασβούργου κτλ. Εμένα με θέλει η ιδέα ε, ότι πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι τα θεσμικά όργανα σε όλα τα κράτη-μέλη ε, και όχι όλα στις Βρυξέλλες, ε, αλλά ας αποφασίσουμε με αέδρα ή εδώ να είμαστε μονίμως στο Στρασβούργο εγώ ή να συνεδριάζουμε μονίμω στι Βρυξέλλε. Αλλά ε, ας σταματήσουμε να σπαταλούμε το χρόνο μα ε, ε, και α εξοικονομήσουμε λίγα χρήματα ε, για τους φορολογούμενους μας. Ο κύριος Γκόλνης, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ε, παρότι υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία στην ψηφοφορία, πρόκειται για μεθόδευση που οτάστε κατά των συνθήκων. Είναι σαφέστατη συνθήκη. 12 ολομέλειε το χρόνο στο Στρασβούργο. Για να καταργήσουμε μία από αυτέ, ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε την, σε μία εβδομάδα δύο συνόδου. Ε, ε, παρακάμπτουμε έτσι τον ερμηνευτικό κανόνα του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, όταν το Κοινοβούλιο θέλησε να περάσει από τι 12 συνόδου στι 11 εδώ και 20 χρόνια βλέπουμε αυτές τις υποχθόνιες μεθοδεύσεις που στόχο έχουν να μην υπάρχει καμία έδρα στο Στρασβούργο και έχουν δίκιο οι συναδελφοί μου. Είναι ανυπόφορη η σημερινή κατάσταση. Δεν χρειάζεται όμως να, γίνει, να γίνουν οι Βρυξέλλες, η Washington DC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας συγκεντρώσουμε όλες τις δραστηριότητε στο Στρασβούργο. Αλλά εδώ ε, χρειάζεται κάτι παραπάνω από τις συνεχίζει σε απόπειρε ε, των γαλλικών κυβερνητικών αρχών. Ο κύριος Πόσελτ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα δεν νίκησε η ομάδα των Βρυξελών την ομάδα του Στρασβούργου γιατί ε, και τι συνεδριάσεις Βρυξέλλες μειώσαμε κατά μία. Άρα δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ε, Βρυξέλλες-Στρασβούργα 1-1. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, εκείνο το οποίο κάναμε είναι ότι ψηφίσαμε αγνώντας το δίκαιο. Η Ολομέλεια του Αυγούστου και του Οκτωβρίου να γίνονται σε μία και μόνο εβδομάδα, αυτό είναι παράνομο. Διότι πρόκειται για Ολομέλειες μία φορά το μήνα όπως αναφέρεται στη συνθήκη. Και πρέπει να πω ότι αυτό δεν εξηγείται με εξοικονόμηση κόστους γιατί τα 70 εκατομμύρια που είναι το κόστος, ε, υψηλό κόστος, το κόστος αυτό δεν προκαλείται από το Στρασβούργο αλλά προκαλείται από το ότι παραβιάζοντας ε, τις ε, συνθήκες ε, συνεχώς πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες αν όμως εστιάσουμε τις εργασίες μας εδώ στο Στρασβούργο θα εξοικονομήσουμε χρήματα και θα έχουμε και ένα μόνιμο δημοκρατικό πρόσωπο της Ευρώπης. Κύριος Βαντάλεν. Είναι εδώ. Ο κύριος Γιάρ, για ένα λεπτό.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζήτησα το λόγο για τις διαπραγματεύσεις για τον προπολισμό γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιμετωπίζεται πάντα με δίκαιο τρόπο. Εμείς ως Ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου είμαστε υπέρ της εξοικονόμησης δαπανών αλλά εξίσου σημαντικό είναι να κάνουμε και σωστά τη δουλειά μας. Ε, το να αυξηθεί λοιπόν η γραμμή του προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό είναι σωστό αλλά η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό αυτό δεν είναι σωστό. Ε, μην ξεχνάτε ότι θα επεκταθούμε, θα αυξηθούμε κατά 18 περαιτέρω βουλευτέ, ε, θα υπάρξει η χρηματοδότηση τη ένταξη τη Κροατία ε, και θα γίνουν και άλλε επενδύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι σε τελική ανάλυση θα ξεβρεθεί ένα ικανοποιητικό ε, συμβασμό. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην πρόοδο εργασιών όσον αφορά την πρόταση Επιτροπή σχετικά με την αναδιοτύπωση τη οδηγία για τι διαδικασίε. Η κυρία Μαζόνι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, αυτό που ενδιαφέρει είναι να προάγουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα, όπως επίσης και στη διαπραγματεύση για τη Μέση Ανατολή. Η έκθεση για την πορεία των διαπραγματεύσεων ως προς την ένταξη Τουρκίας ε, καθορίζεται και χαρακτηρίζεται από αντίδραση των τουρκικών δυνάμεων απέναντι σε κάποια βασικά στοιχεία της Συμφωνίας Σύνδεσης. Εγώ κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι για λόγους δικαιοσύνης, ελευθερίας ενημέρωσης, θρησκευτική ελευθερία και πολλά άλλα οι ε, τουρκικές αρχές δεν έχουν σημειώσει ε, ε, τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή δεν μπορούν να μας οδηγούν στο να αγνοούμε την ελευθερία βασικών ε, δικαιωμάτων και απόψεων. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, δεν θα πρέπει να παρασύρονται και δεν θα πρέπει να ματαιώσουν τη διμερή σχέση που υπάρχει. Η δική μου ανησυχία είναι ότι αυτή η παραδοχή που αναφέρεται, η υπόθεση για ειδική προτιμησιακή συμφωνία, αυτό ε, θα μπορούσε να καθυστερήσει την ένταξη που θα πρέπει να παραμείνει βασικό μα στόχος. Ευχαριστώ. Κυρία Ζωνή, ε, μιλήσατε για λάθος έκθεση και πάνω από ένα λεπτό. Μετά είναι ε, αυτή η έκθεση για την Τουρκία. Τώρα ασχολούμαστε με την προηγούμενη έκθεση. Όταν φτάσει φτάσει η ώρα της έκθεσης για την Τουρκία θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, αυτές οι περιοχές ε, οι υδάτινες περιοχές έχουν μεγάλη έκταση στην ε, ε, υδρόγειο και κυρίως έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομική ανάπτυξη. Η περιοχή του Ατλαντικού για τις μεταφορές, ε, για την ενέργεια, για την αλληλεία έχει ιδιαίτερη σημασία. 50% του πετρελαίου, του φυσικού αερίου προέρχονται από εκεί καθώς και των αλληλευτικών αποθεμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο καταστροφής μπορεί να είναι οι συνέπειες για τις παράκτιες περιοχές. Χρειαζόμαστε μια ορθή τη για την περιοχή του Ατλαντικού, τόσο ώστε να αναβαθμιστεί η διακυβέρνηση και να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων των περιοχών. Πρόεδρο 2010 για την Τουρκία, πρώτος ο κύριος Καλινόφσκι, για ένα λεπτό. Mr. Kalinowski, one minute on Turkey. Κύριε Καλινόφσκι, ένα λεπτό έχετε για την Τουρκία. Panie Przewodniczący, jakaś pomyłka. Ja mam zabrać głos w polityce przemysłu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα πρόκειται για λάθος. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Συγγνώμη, Πρόεδρε, ε, προφανώς υπάρχει λάθος. Ε, ήθελα να πάρω το λόγο για να μιλήσω για την βιομηχανική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Είσαστε και στον κατάλογο της Τουρκίας όμως. Ε, η κυρία Μαζόνη. Ε, συγγνώμη πρόεδρε, τώρα τι να κάνω, ε, να μιλήσω τώρα για την ε, Ατλαντική Στρατηγική. Ε, μάλιστα, μάλιστα, γιατί να μιλήσετε. Εντάξει, ε, πρόεδρος, ε, δεν είναι δικό μου λάθος ε, που δεν ακούσατε για ποια έκθεση κληθήκατε να μιλήσετε. Μιλήσατε πριν για την επόμενη, τώρα πάτε για την προηγούμενη. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω για την Ατλαντική Στρατηγική, αλλά προηγουμένω μου δώσετε το λόγο να μιλήσω για την Τουρκία. Τέσπα. πρόεδρε. Συγγνώμη, πρόεδρε, αποσυντονίστηκα. Λοιπόν, το ψήφισμα αυτό πρέπει να το εντάξουμε στο πλαίσιο της ε, οδηγίας του 2008, την ε, στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως ακριβώς είπε και ο συνάδελφος που παρενέβη προηγουμένως, ε, το πλαίσιο είναι της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γιατί αυτή η οδηγία καθορίζει κοινέ αρχές και με βάση αυτό τα κράτη-μέλη μπορούν να επεξεργαστούν τη δική τους στρατηγική σε συνεργασία και με τρίτες χώρες για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική κατάσταση σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθεί η στρατηγική για τον Ατλαντικό και με βάση ε, τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου του περασμένου Ιουνίου. Το ψήφισμα λοιπόν που κατατέθηκε ε, ξεπερνάει αυτό το πλαίσιο και προτείνει ε, αυτά τα οποία παρουσίασε η Επιτροπή, δηλαδή μια στρατηγική που να μην είναι απλά και μόνο ε, σχετική με το θαλάσσιο περιβάλλον. Εγώ λοιπόν εύχομαι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή θα λάβει υπόψη αυτά που ελέγχθησαν εδώ και έτσι θα καθορίσει μια νέα ε, στρατηγική ε, για το θαλάσσιο περιβάλλον και γι' αυτό λοιπόν εγώ δήλωσα αποχή Πρόεδρε. Ε, πίσω το θέμα της Τουρκίας τώρα η κυρία ε, Σκριτλεύσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, με ικανοποίησε η έκβαση της ψηφοφορίας για την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Είμαι πεπισμένη ότι οποιοδήποτε διάβημα αποσκοπεί στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων αξιών αξίζει να τύχει της υποστήριξής μας. τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η Ένωση οφείλουν να συνδράμουν την Τουρκία στις προσπάθειες που καταβάλει ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα βασικότερα θέματα, ελευθεροτυπία, δικαιώματα των γυναικών, προστασία των ε, εθνικών μειονοτήτων κτλ. Επίσης, για το επιπρόσθετο πρωτόκολλο για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας θα πρέπει να προχωρήσουν εργασίες. Για ένα λεπτό.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 Κύριε Πρόεδρε, εγώ τάχθηκα υπέρ του ψηφίσματος για την Τουρκία γιατί η συνταγματική μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα στις 12 ε, Σεπτεμβρίου αναγνωρίστηκε ομόφωνα ως ένα σημαντικό βήμα από την Τουρκία προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. Βεβαίως η Τουρκία πρέπει να κάνει ακόμα πολλά βήματα και ε, ανησυχώ για την ε, σύλληψη των δημοσιογράφων. Η Τουρκία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βεβαίω σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας οι εμπορικές ανταλλαγές ε, ε, βοήθησαν στο να γνωριστούν οι λαοί ειρηνικά ε, θεωρώ ότι μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω βήματα στη σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσα από τη θάλασσα, από την Αδριατική, το Τυρινικό πέλαγος. Εξίσου σημαντικέ ε, είναι και η ε, ε, συνδρομική διασύνδεση. Με τον τρόπο αυτό, με αυτέ τι διασυνδέσει, μπορέσαμε να βελτιώσουμε τι εμπορικέ συναλλαγέ και θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η έκθεση για το 2010 που κατατέθηκε δείχνει ότι έχουν ε, ε, υλοποιηθεί βαθύτατες αλλαγές ε, στη χώρα αυτή. Κυρίως έχουν γίνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που εκδημοκρατίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή στην Τουρκία. Όμως θα θέλαμε να συμβιωθεί ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο σε κάποιους τομείς. Είναι σημαντικό ε, να δούμε τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες ε, και δεν μιλώ μόνο για το κυπριακό ζήτημα γιατί δεν έχουν ακόμη καταλήξει διαπραγματεύσεις ε, μιλώ κυρίως για, τις, για τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ελπίζω ότι με την έκθεση αυτή, μετά την έκθεση αυτή θα σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στην Τουρκία ούτως ώστε η χώρα αυτή να γνωρίσει αλλαγές όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα αλλά και σε άλλους σημαντικότερου τομεί, δηλαδή στον τομέα των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Είμαι ε, σίγουρο σχεδόν ότι ο κύριο Μπίμπ ε, μίλησε και όχι ο κύριο Μπίν Ε, δίκαιο έχω. Μπίλεν τώρα λοιπόν. Ο κύριο Μπίλεν θα πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επειδή μετέχω στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία ΕΕ Τουρκίας, γνωρίζω αυτά τα ζητήματα και πιστεύω ότι το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών, του δικαστικού συστήματος, το θέμα της ελευθερίας των μαζικής ενημέρωσης, του θέμα των ενόπλων δυνάμεων. Ε, είναι όλα σημαντικότατα ζητήματα και πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Ε, και κυρίω πρέπει να μεταρρυθμιστεί ε, το εκλογικό σύστημα. Άλλο ε, πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι η φόνη τιμή και η ενδοοικογενειακή βία. Επίσης το θέμα της, των συνόρων με την Αρμενία, το θέμα της Κύπρου, άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν και εμείς θα πρέπει να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολωνίας φυσικά. Σας ευχαριστώ. Ο Ποητό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας ε, δήλωσε αποχή, όχι γιατί δεν συμφωνώ με την ανάλυση ε, και παρότι υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, εξακολουθεί να υπάρχει λογοκρισία Νομίζω αυτό και από μόνο του λέει πάρα πολλά και εγώ δήλωσα αποχή κυρίως ε, γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να ζητήσει πολύ αυστηρότερα μέτρα. Εάν η Τουρκία αρνείται να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις ε, τότε και εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευόμεθα την ένταξή της. Έχει φτάσει πια η στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει την πλήρη ανάκληση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. <coughs> <coughs> Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι υπήρξε κάποια πρόοδος στην Τουρκία κατά τα τελευταία έτη, αλλά αν δούμε λιγάκι τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης που έχουμε για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ. Και θέλω να πω ότι ε, όσο ζω εγώ δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Τουρκία είναι τόσο μακριά από τα ε, δικαιώματα των ανθρώπων, των ε, γυναικών και των παιδιών που είναι θεμελιώδης αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, εξάλλου είναι σημαντικό να μην αγνοούμε και την κατάσταση στην Κύπρο. Όσο η Τουρκία έχει υπό την κατοχή της το ίμιση του εδάφους ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωσης πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Δεν μπορούμε να δεχόμεθα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόζει τώρα η Τουρκία. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να μετακινηθούν προς την δημοκρατία αλλά πρέπει να τους πούμε και με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αντρανίσει. Κύριε Πρόεδρε, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία ε, θα κριθεί ως, ε, κάποια στιγμή ως ε, κολοσιαίο λάθος. Εμείς ε, δείξαμε καλή θέληση, αλλά θα έπρεπε ευθύ εξ αρχή να πούμε, κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένταξη, ας βρούμε κάποια εναλλακτική λύση. Και αντί να το κάνουμε αυτό, εμείς τους αφήσαμε να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβήκαμε σε υποσχέσεις που δεν θέλουμε να τις ε, εκπληρώσουμε. Ελάτε όμως στη θέση της ε, Άγκυρας, κάνανε κάποιες παραχωρήσεις και στην Κύπρο. Βέβαια οι Τουρκοκύπροι τάχτηκαν υπέρ της ε, στην ε, Κύπρο, το απέριψαν οι Ελληνοκύπροι. Ε, τους επιβάλαμε πάρα πολλά πράγματα και τελικά θα τους κοροϊδέψουμε και γι' αυτό λοιπόν κινδυνεύουμε να επιτύχουμε αυτό που δεν θέλαμε, το να υπάρχει μια εχθρική στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε παρελθόν δεν πρέπει να επαναληφθεί και στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, παρότι συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις του Ντέλφου Μπίπερτ, εγώ υπερψήφισα την έκθεση, γιατί για άλλη μια φορά λέμε με απόλυτη σαφήνεια στην αρχή της έκθεσης ότι για μας οι διαπραγματεύσεις είναι μια μακρά διαδικασία με, ανοιχτό, με ανοιχτή έκβαση. Εμείς απορρίψαμε την πρόταση των Πρασίνων που θέλησαν να μας δεσμεύσουν ε, για πλήρη ένταξη. Ε, αυτό το έκαναν και οι σοσιαλδημοκράτες υπέβαλαν σχετική πρόταση. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα και να πούμε με απόλυτη ειλοκρίνεια στου ε, Τουρκου, όπω είπε και ο κ. Μπίπερτ, ότι πλήρη ένταξη τη Τουρκία δεν τίθεται καν τέτοιο θέμα, γιατί αυτό θα ξεπερνούσε την Τουρκία ε, και θα ε, έφερνε και στα όρια τη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικά ενοποιημένη Ευρώπη με μέλο στην Τουρκία, αυτό είναι αδύνατο και αυτό είναι ψέμα που πρέπει επιπλέον να το εγκαταλείψουμε. Και όσον αφορά την πρόοδο, αυτή είναι προ όφελο τη ίδια τη Τουρκία που είναι μέλο ε, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δικό μα στενό σύμμαχο. ja bym chciał tu nawiązać do dyskusji która się toczyła na tej sali. Κύριε Πρόεδρε, κατόπιν ε, Συζήτηση για την προσχώρηση του Μαυρογονίου έθεσα την ερώτηση στους της Κομισιόν και Συμβουλίου τι χρονοδιάγραμμα προβλέπουν για τη σχετική διαδικασία. Πότε το Μαυροβούνιο θα θεωρηθεί χώρα υποψηφία. Δεν μου απήντησαν εγώ ψήφισα υπέρ του κειμένου. Άλλωστε είναι κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Κροατία. Ψήφισα υπέρ και για αυτό το λόγο. Επίσης αυτό το κείμενο από τη λέμε καθηγητήρια γραμμή ούτως υπήρχε και για άλλες βαλκανικές χώρες. Επίσης ψήφισα υπέρ διότι κατά τρίτον είναι το κείμενο αυτό ένα κείμενο σημαντικό που αποδεικνύει κάποιες ε, θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε την πολιτική διεύρυνση να την εντάξουμε μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Και όπως προβλέπετε, μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία και εν συνεχεία η Κροατία το φθινόπωρο με τη δική μας ε, την ψήφο ε, να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Κροατία θα πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο το μεθεπόμενο χρόνο. Και μετά πρέπει να συνεχιστεί η πορεία. Δηλαδή πρέπει να εντάξουμε και τις άλλες χώρες πρώτα, τη Μακεδονία και μετά το Μαυροβούνι και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις άλλες χώρες της ε, περιοχής ότι εφόσον ε, πληρούν τα κριτήρια έχουν θέση εδώ γιατί αντίθετα με την Τουρκία αυτές είναι ευρωπαϊκές χώρες που είναι αυτονόητο ότι έχουν μέλλον στη δική μας την οικογένεια. Ειδικά το Μαυροβούνι είναι μια μικρή χώρα με μια μακρά ευρωπαϊκή ιστορία και ήδη χαίρομαι πάρα πολύ για τις διαπραγματεύσεις με

Πρόεδρε, ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά στον αγώνα κατά τη διακριτική μεταχείριση στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν συμφωνώ με την εισηγήτριά μα που ισχυρίζεται ότι όσον αφορά ε, στη διακριτική μεταχείριση εθνοτικών μειονοτήτων, αυτή μπορεί να περιοριστεί. Ο κοινωνικό αποκλεισμό των Ρωμά εξακολουθεί να υφίσταται και παραμένει μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ειδικοί και συγκεκριμένοι παράγοντες, ε, ε, γεωγραφικά μειονεκτήματα, ε, κατάρρευση της οικονομίας, της κατευθυνόμενης οικονομίας. Όλα αυτά οδήγησαν στον περισσότερο εντονότερο αποκλεισμό τους. Και υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Πρέπει λοιπόν να τους εντάξουμε. Ένα μεγάλο τμήμα των Ρωμά βρίσκονται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη κατάσταση που τα μέτρα που προβλέπονται για, τον, για την ένταξή τους ε, δεν αρκούν, ε, δείχνουν πάρα πολλά ε, κενά, κυρίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Συζητούμε εδώ για τους Ρωμά στο Κοινοβούλιο και λέει μια πολιτική ομάδα ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Άλλες πολιτικές ομάδες πάλι λένε ότι ε, δεν θα πρέπει να σπαταλούμε κονδύλια για την ε, στρατηγική ε, των Ρωμά, γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες. Τέλο πάντων, παρά την ε, διχογνωμία, η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα είναι καλή. Ε, και αυτό που πρέπει να κρίνουμε είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει δαπανίσει πολλά κονδύλια για την ενσωμάτωση των Ρωμα. Πρέπει να δούμε ποια προγράμματα προήγαγαν ε, την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων και να εκπονήσουμε μία πραγματική, πραγματικά αποτελεσματική πολιτική και άρα ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση αυτή η έκθεση. Για ένα λεπτό. Sì, grazie. Presidente, con l'approvazione odierna della relazione di iniziativa το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα προς την κατεύθυνση της ε, πραγματικής ένταξης ε, των ε, Ρωμά. Η περιθωριοποίηση των Ρωμά θα πρέπει να έρθει να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και να υπάρξει και προστασία των ευαίσθητων κατηγοριών. Εμείς θεωρούμε ότι πολύ σωστή, πρέπει, σωστή είναι και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση στο κείμενο προβλέπονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να εγγυηθούν τη σωστή χρήση των προβλεπόμενων κονδυλίων. Πάνω απ' όλα μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους ε, γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ανάληψη ευθυνών απέναντι στους Ρωμά έτσι ώστε να είναι και αποτελεσματική η ενσωμάτωσή τους. λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά ε, και δεν θα πρέπει ε, να υποτιμούμε τις διακρίσεις εις βάρος τους. Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, ε, δεν μπορεί να μην υπάρχει νομιμότητα. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν ε, σε πολύ κακές συνθήκες, ε, είναι παράνομοι πολλές φορές, ε, καταλήγουν και προβαίνουν σε ληστείες, σε κακοποίηση των παιδιών. Είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν στο χώρο της εργασίας. Αυτή λοιπόν είναι πραγματικότητα πολλών κοινοτητών Ρωμά και στη δική μου τη χώρα και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν είναι υποκριτικό να ισχυριζόμεθα ότι η ευθύνη βρίσκεται μόνο σε επίπεδο θεσμών και όχι σε επίπεδο εκείνων που έχει μετακυλήσει το βάρος στον Ρωμά στις πλάτες όλων των πολιτών. Πρέπει να υπάρξει σωστή εφαρμογή της Οδηγίας 38 του 2004 που προβλέπει αυστηρές προδιαγραφές ε, για την παραμονή μιας κοινότητα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Για όλους αυτούς τους λόγους εγώ ε, δήλωσα αποχή. Ένα λεπτό. Grazie, <clears throat> Presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση της ε, συναδέλφου Γιωράκ, Γιαρούκα υποβάλλεται σε μια στιγμή κατά την οποία ε, καθορίζεται η βάση και για τις μελλοντικές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, Ρωμά. Ε, εκείνο που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα στηθεί σε 7 και 8 Απριλίου. Υπάρχουν λοιπόν ελάχιστες προδιαγραφές δεσμευτικέ στον τομέα της παιδείας, της απασχόλησης, της στέγασης και των υγειονομικών συνθήκων. Μεγαλύτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να ενταχθεί η μειονότητα των Ρωμά εκεί εκείνο το οποίο συμμερίζομαι, αποκινούμε άλλες χώρες, είναι ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τον ε, ρόλο της, ε, του, του, του καθοδηγητή όσον αφορά κυρίως ε, την συμπερίληψη των Ρωμά. Οι Ρωμά βέβαια και αυτοί οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τις υποχρεώσεις. Κροτσέτα, παρακαλώ. Δεν είναι εδώ ο κύριος Κορτσέτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας υποστήριξε την έκθεση αυτή, διότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση ε, ε, και καλεί έναν οδικό χάρτη και μια ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρωμά. Βασίζεται στην, στις, στα στοιχεία που υπάρχουν και σχετικά με τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων Ρωμά μέσα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα προβλέπει ελάχιστα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εκπονηθεί μια πραγματική πολιτική ενσωμάτωση. Ε, η στρατηγική αυτή καλύπτει όλο τον ειδών τη παραβία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Ρωμά. Ε, καλή, αποτελεσματική, ε, καλή, αποτελεί συγγνώμη, έκκληση για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των Ρωμά και η πολιτική μου ομάδα εκτιμά ιδιαίτερα αυτά που προβλέπονται για τα παιδιά των Ρωμά για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση στα σχολεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση πρωτοβουλία και δείχνει την ανάγκη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ε, κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση των Ρωμά που αυξήθηκε μετά την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Θα πρέπει να έχουμε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο και να αποφύγουμε την αντιμετώπιση αυτού του θέματος με προαιρετικές μόνο και οικειοθελείς διατάξεις γιατί είναι ανεπαρκείς και δεν εξυπηρετούν το στόχο μας. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ως μόνιμο όργανο την Task Force για τους Ρωμά και ένα αντίστοιχο μηχανισμό που έχουμε για την αξιολόγηση της εσωτερικής αγοράς να προβλέψουμε και για τους Ρωμά. Τέλος, η Ευρώπη θα πρέπει να μην φυστεί προσπαθειών για να ε, εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών της, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων και την, ε, το σεβασμό όλων των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνική ένταξη στο Ρωμά είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε να ενταχθούν οι Ρωμά στην κοινωνία και να μην μείνουν εγκλωβισμένοι στη δική τους πραγματικότητα, με σεβασμό όμω της πολιτικής πραγματικότητας και της κοινωνική στην οποία ζουν. Ο κύριος Αντινόρο. Με τη σημερινή ψηφοφορία δώσαμε μια νέα όθηση για την οριστική λύση του προβλήματος, αλλά δεν νομίζω ότι επιλέξαμε την καλύτερη δυνατή λύση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι άνω των 300 τροπολογιών που υποβλήθηκαν ε, μετατράπηκαν σε 28 συμβαστικές τροπολογίες που εγκρίθηκαν όλες και καθορίζουν καλύτερα τη στρατηγική και τους στόχους της ε, στρατηγικής αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μόνιμη Task Force θα πρέπει να εξασφαλίσει την συμπερίληψη των στοιχείων αυτών και τα κράτη-μέλη να ορίσουν έναν υψηλό βαθμό, ελπίζουμε, υπάλληλο που θα διαδραματίσει το ρόλο αξιωματούχου επαφής για τη στρατηγική αυτή. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο φιλόδοξοι στην έκθεσή μας αν είχαμε στείλει και κάποια μηνύματα για τους ε, Ρωμά και τις υποχρεώσεις και δικαιώματά τους και στη χώρα ε, υποδοχής. Έτσι θα προβλέπαμε καλύτερη συνύπαρξη των ε, Ρωμά στις κοινωνίες που διαβιώνει. κυρία Αντζελίλη. Έχουμε πολλά παιδιά δυστυχώ που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση. Δεν θέλουμε πια τέτοια φαινόμενα και η έκθεση για Ρούκα προσπαθεί να καταπολεμήσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Πέραν της διακήρυξης αξιών, περιμένουμε και την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τον Απρίλιο, ώστε να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη και καλύτερο συντονισμό σε ό,τι αφορά την πολιτική των Ρωμά. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους της τα κοινοτικά κονδύλια, ώστε οι τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν κυρίως αυτά τα προβλήματα να έχουν καλύτερα εφόδια για να τα αντιμετωπίσουν. Θέλουμε ιδιαίτερες διατάξεις για την εργασία, ε, την υγεία, θέματα διασπαραμονής. Η οδηγία όμως έχει και κάποια κενά. Γιατί τι θα γίνει με τις κυρώσεις σε περίπτωση που δεν γίνουν σεβαστές αυτές οι διατάξεις. Υπάρχει ένα κενό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γιαρόκα για την εξαιρετική εργασία που έχει κάνει, συνοψίζοντα επίσης ε, τις διάφορες θέσει των Ευρωβουλευτών και θέτοντα του πραγματικού στόχου τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρωμά, για την καταπολέμηση τη διακριτική μεταχείρισης, καθώ επίση και την εξασφάλιση τη παροχή ε, ε, κατάλληλων υπηρεσιών προς ανθρώπου αυτού, καθώ επίση και του κατάλληλου επίπεδου εκπαίδευση, παιδεία και στέγαση. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε πραγματικά την ένταξη των Ρωμά, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και μέσω τη τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει όμω εδώ πέρα η απαραίτητη επίβλεψη της διαχείρισης του όλου συστήματος προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όντω όλοι οι Ρωμά θα ενσωματωθούν στο σύστημα αυτό. Τι θα γίνει όμως με τους ε, Ρωμά εκείνου οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν στο σύστημα, τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένω να μην καταφέρουν να υποβληθούν στα συστήματα πρόνοια τα οποία εμεί προτείνουμε. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πήρα το λόγο και προηγουμένως για την έκθεση αυτή και για το περίπλοκο αυτό ζήτημα. Πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους και ιδεώδη που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί παράδοση των ανθρώπων αυτών να μετακινούνται πάρα πολύ. Και στη δική μου τη χώρα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό Ρωμά Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς και καλύτερη πληροφόρηση προς τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα μέσα, νομοθετικά μέσα, τα οποία να λειτουργούν σωστά και κάθε κράτος μέλος πιστεύω φέρει μια πολύ σημαντική ευθύνη για την ένταξη των Ρωμά. Ο κύριος Μικολάσης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, εδώ μιλάμε για το θέμα τη ένταξη της ένταξης των Ρωμά. Οι Ρωμά ζουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και σε δυτικέ και σε ανατολικέ χώρες και πρέπει να διαπιστώσουμε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στι χώρες τη Δύση Εδώ και πολλά χρόνια, χάρη στη δημοκρατία, οι όροι και οι συνθήκες συνεχώς βελτιώνονταν. Στη χώρα μου, στη γειτονική μας χώρα, στην Ουγγαρία, γνωρίζουμε τα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία πολλές φορές είναι παρόμοια με προβλήματα που υπάρχουν και στη Δύση. Και συχνά για το θέμα της ένταξης, Λέμε ότι είναι σημαντικό να επιτύχει ένταξη στην αγορά εργασίας και ότι ε, ο πληθυσμός αυτός θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην εργασία, πρόσβαση στην ε, παροχή υγείας, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτά είναι σημαντικές απαιτήσει που πρέπει να φροντίσουμε. Ευχαριστώ. Tämä Livia Jarokan Ευχαριστώ. Η έκθεση Γιάροκα είναι σημαντική έκθεση και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι καταλαβαίνουμε ότι έχει φτάσει πια η εποχή που πρέπει να αρχίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασχολούμαστε με το θέμα. Όλοι πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει για του Ρωμά. Δεν αρκεί όμως να έχουμε μια καλή έκθεση, χρειαζόμαστε και δράση για τα θέματα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον για να διασφαλίσουμε ότι η έκθεση αυτή δεν θα παραμείνει απλώς ε, ένα ευχολόγιο, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση για τους Ρωμά βελτιώνεται αισθητά στο, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης πρέπει να υπάρξει και κάποια συνέχεια στην έκθεση αυτή. Ενδεχομένως να ορίσουμε κάποιον εκπρόσωπο, ο οποίος θα εξετάσει πώς μπορεί να μεταφερθεί στην πράξη αυτή η έκθεση. Πρώτος ο κύριος Μαστέλα για ένα λεπτό. E Ευχαριστώ. Η πρόσφατη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση χτύπησε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ανέδειξε τη σημασία της για την ευρωπαϊκή οικονομία. Βέβαια, επικεντρωθήκαμε στο γεγονό τη αυτορύθμιση των αγορών και αυτό γίνεται μέσω κάποιων μεμονωμένων μέτρων χωρίς όμως κανένα συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 για πρώτη φορά αναγνωρίζει την ανάγκη μιας νέα προσέγγισης. Έχει και η ώρα επιτέλους να, να αξιοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλε τι δυνατότητε που έχουμε για να αναπτύξουμε τη βιομηχανική μας βάση η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να κρατήσει τον ηγετικό της ρόλο σε νευραλγικούς τομείς. Και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλέξει το, ρόλο, το μέλλον της, θα πρέπει να φροντίσει και μια για μια καλύτερη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για έναν καλύτερο συντονισμό, ώστε να υλοποιήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της απασχόλησης μέσω της φορολογικής αναρμόνισης και του φόρου στις εταιρείες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση Λάγκε ασχολείται με ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ και τα οποία γίνονται ακόμα πιο σημαντικά στα πλαίσια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης που έχει πειράσει πολύ αρνητικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θεωρώ ότι το μήνυμα το οποίο δίδεται από την έκθεση είναι ιδιαίτερα θετικό καταφέρνει η έκθεση αυτή να αφαιρθεί σε όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου να καταφέρουμε να διηγηθούμε σε μια οικονομική ανάκαμψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το κατάλληλο επίπεδο έρευνα και επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, προκειμένου να καταφέρουμε να τονώσουμε το, την βιομηχανία, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μάλιστα στι φιλοδοξίε τη η έκθεση ξεπερνά και του αρχικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε υπόψη τι τροπολογίε μα, τι προτάσει μα. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης που θέτει πλέον συγκεκριμένους στόχους και που ε, θέτει επίση κάποια μοντέλα επίβλεψης τα οποία είναι τόσο από τα πάνω προς τα κάτω όσο και από τη βάση προς τα πάνω. Θα πρέπει να υπερψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση αυτή που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα θετική. Δεν εδώ. Ο κύριος Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική. Ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ε, απασχολούν και κάποιες ευρωπαϊκές, ε, εθνικές με ενώσεις βιομηχανών. Ωστόσο θα έπρεπε να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις, κάποια ζητήματα τα οποία δεν διευθετούνται στην έκθεση αυτή, όπως για παράδειγμα νέα νομοθετικά μέτρα όσον αφορά την ενέργεια και την επάρκεια των ενεργειακών πηγών. Επίση, πρέπει να μα απασχολήσει και το ζήτημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και θα πρέπει να μας απασχολήσει επίση και το ζήτημα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί πιστεύω ότι ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά όργανα να καταρρύψουν όλα τα εμπόδια τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή προκειμένου να εφαρμοστεί το φιλόδοξο αυτό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Καλινόφσκι. Φυσικά η βιομηχανία στον κόσμο αναπτύσσεται με ραγδαίου ρυθμούς. Για να μην μείνουμε πολύ πίσω από την Κίνα και την Ινδία, χρειαζόμαστε άμεσες αλλαγές. Θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι περισσότερο στον κόσμο από τις ε, βιομηχανίες που μετακατίστανται. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη φαρμακολογία, στην επιστήμη και στι καινοτόμε ενέργειες, ακόμη και στο γεωργικό τομέα. Δεν ε, χρειαζόμαστε λοιπόν νέες, νέες διατάξεις που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που θα σέβονται το περιβάλλον, θα είναι υγιεινά και φυσικά θα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέτοια χρειαζόμαστε σε μια νέα κοινωνία και φυσικά χρειαζόμαστε ε, καινοτόμες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις δημογραφικές αλλαγές και στον γυράσκοντα ευρωπαϊκό πληθυσμό. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η βιομηχανική πολιτική είναι συστατικό τμήμα της ε, οικονομικής πολιτικής και θα πρέπει να προωθήσουμε μια αηφόρο ανάπτυξη και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πεδίο έντονου ανταγωνισμού και γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει ενεργό πολιτική για να προφυλάξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να την οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της οικονομίας παράλληλα. Αυτό θα πρέπει να το διασφαλίσουμε θεσπίζοντας τους κατάλληλους όρους μέσω των συμβάσεων, μέσω του δικαίου του παραγωγού και μέσω ε, των δικαιωμάτων που θα διασφαλίζουν τη βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να παράσχει πλεονεκτήματα ανταγωνισμού και στους ανθρωπίνους πόρους και αυτό εξαρτάται και από τις επενδύσεις στην οικονομία. Ευχαριστώ. έχουμε με ε, πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία, τρία τέταρτα των προϊόντων μας ε, τα εξάγουμε. Η βιομηχανία έχει τεράστιο τεράστια σημασία για την οικονομία μας, απασχολεί πολύ ε, μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αλλά δεδομένου του πολύ ε, σημαντικού παγκόσμιου ανταγωνισμού θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τη συστηματική της ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020 είναι μια απόπειρα μιας νέας προσέγγισης που θα αξιοποιεί καλύτερα τις δυνατότητες που μας δίνει ο εξυγχρονισμός της ε, βιομηχανικής βάσης στα κράτη-μέλη θα πρέπει ταυτόχρονα βέβαια να εξασφαλίσουμε και τις ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Έτσι δημιουργούμε ε, τις προϋποθέσεις για να κρατήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Επίση, ε, πολύ, πολύ υποσχόμενη είναι μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα ε, περάσει από την, ε, από την έμφαση στην παραγωγή στην έμφαση στην επιστήμη και στην επιστημονική γνώση. Είμαι υπέρ της έκθεσης του κ. Μπέρντ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε εδώ πέρα για έναν τομέα ο οποίος ε, εκπροσωπεί 57 εκατομμύρια εργαζομένους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα εξαγωγών, αντιστοιχεί στο 1 τρίτο του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Επομένως, χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη ξεχωριστή τομεακή πολιτική για την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Χρειαζόμαστε προφανώς μια βιομηχανική δραστηριότητα, ιδιαίτερα καινοτόμα, προκειμένου να καταφέρουμε να μείνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου και προκειμένου να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα προστατεύει και το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου ιδίως στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις εμπορικές που θα κάνουμε, για να καταφέρουμε να προασπίσουμε τον βιομηχανικό μας τομέα, καθώς επίσης και τις θέσεις απασχόλησης τομέα αυτού. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να θέσουμε σε πρώτη γραμμή ως βασική προτεραιότητα την πραγματική οικονομία και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε και τα φαινόμενα κερδοσκοπία Oh. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μια τέτοια έκθεση. Θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχουν κρίσεις, αλλά ακόμα χειρότερα θα ήταν το να μην μαθαίνουμε και να μην διδασκόμαστε από τις κρίσεις. Νομίζω ότι από την τελευταία κρίση διδασκόμαστε πράγματα και για τη βιομηχανική πολιτική και ξέρουμε ότι και πριν από την κρίση υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που ε, μπορεί να θεωρούσαν ότι ε, η οικονομία μπορεί να αποτελέσει μόνο πηγή ε, εξοικονόμησης πόρων. Νομίζω ότι με την κρίση μας δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούμε με την βιομηχανική πολιτική, με την αηφόρο ανάπτυξη, με το μέλλον της βιομηχανικής πολιτικής, με την καινοτομία και την επιστήμη και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε την έκθεση αυτή και ελπίζω να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στο μέλλον περαιτέρω. Ευχαριστώ. Κέλλη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ αυτής ε, της έκθεσης, την οποία θεωρώ ε, καλή και νομίζω ότι ήταν ο καιρός, ε, έφτασε ο καιρός να ασχοληθούμε με τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια εμείς καθυστερήσαμε σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες και ελπίζω στο μέλλον αυτό να διορθωθεί. Θέλω να εκφράσω μια ανησυχία για ένα σημείο στην αιτιολογική έκθεση στη σελίδα 32, εκεί που ζητά την εναρμόνιση των, της εταιρικής φορολογίας. Η χώρα μου δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Ο εταιρικό φόρο, ο φόρο τη εταιρεία είναι για μα πολύ σημαντικό θέμα και κάθε χώρα θα πρέπει να θεσπίζει τα δικά τη ποσοστά. Είναι γνωστό ότι ορισμένε χώρε έχουν υψηλό εταιρικό φόρο, αλλά στην πραγματικότητα καταβάλλονται λιγότερα χρήματα. με χαρά ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα που αποτέλεσε το καρπό μιας συζήτησης για την πραγματική οικονομία έγινε δεκτό με μεγάλη πλειοψηφία. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις ε, που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση για την βιομηχανική πολιτική και την πραγματική ε, ευρηματικότητα και δημιουργικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 που προσπαθεί να αναχαιτήσει το φαινόμενο της μετακατάστασης και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Και σίγουρα στο πλαίσιο αυτό η βιομηχανική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο και του σχετικού ψηφίσματος. Μπορούμε να χάσουμε στην Ευρώπη την παραδοσιακή μας βιομηχανία. Όχι, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Έτσι ε, φάνηκε και στη συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης ε, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις πρώτες ύλε και στις ενεργειακές πρώτες ύλε. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία με την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιστήμη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια και στις διάφορες πολιτικές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνδυάσουμε τη γεωρική πολιτική με τη βιομηχανική αλλά και την εμπορική πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί και να υποστηρίξει στεναρά τη βιομηχανική πολιτική, να αντιμετωπίσει το κίνδυνο από την κρίση, την ανταγωνιστικότητα των ε, τρίτων χωρών και την, ε, την υποστήριξη από το τρίτο πρόγραμμα πλαίσιο γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε την ιδιωτική επένδυση και να ε, ευνοήσουμε τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Έτσι θα δημιουργήσουμε ειδικευμένε θέσει εργασίας, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε και, το επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό των περιφερειών που έχουν αναπτύξει κάποια δίκτυα καινοτομία και κάποιου πόλου έλξη και αριστεία, τα κλάστερ. Αυτό συνέβη στο Εοσκάδη, στη χώρα των Βάσκων. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τη γνώση των περιφερειών. α μην στρέψουμε την πλάτη μα σε αυτή την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τόσε απειλέ ε, αυτή τη στιγμή που η αναγνώριση των περιφερειών θα μα επιτρέψει να ε, δώσουμε και να κατοχυρώσουμε την ηγετικό μα ρόλο στη βιομηχανική πολιτική. Δεν είναι εδώ ο Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτη συνεδρίαση ω στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you.